Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε την επανέναρξη της ε, συζήτησης. Υπάρχουν ε, τα πρακτικά της χθεσινής ε, συνεδρίασης. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, άρα...